Good morning, Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας συνεδρίαση. Πρωτού ξεκινήσουμε επίσημα με τη συνεδρίαση, θα ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Καταρχάς, χρησιμοποιήστε παρακαλώ πολύ τα ακουστικά σας, γιατί θα μιλήσω στη γλώσσα μου, τα τσέχικα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η συνεδρίασή μας μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Σήμερα συνεχίζουμε τη συνεδρίαση την οποία ξεκινήσαμε χθες. Θα περάσουμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, παρουσίαση μελέτης για τη διάδοση των πυρηνικών όπλων στη Βορειοανατολική Ασία. Η μελέτη αυτή αναφέρεται στις προκλήσεις της πυρηνικής πολιτικής της Βορείου Κορέας, και αναφέρεται επίσης στις επιπτώσεις που πολιτική αυτή θα μπορούσε να έχει για το καθεστώς μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Η δική μας υποεπιτροπή ζήτησε την εκπόνηση μιας μελέτης από κοινού με την αντιπροσωπή για τις σχέσεις με την Κορατική Χερσόνησο. Θα παρουσιάσει τη μελέτη αυτή ο συγγραφέας της, ο συντάκτη της, ο κύριος Μπενζαμά Ότ Κουβερτούρα, ο οποίος εργάζεται στο Ίδρυμα Στρατηγικών Μελετών του, Παρισιού. Σας δίνω λοιπόν το λόγο. Thank you very much, Mr. President. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματική τιμή να βρίσκομαι σήμερα το πρωί εδώ πέρα, στη δική σας συνεδρίαση σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συζητήσω μαζί σας κάποια στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι αποτελούν πρόκληση για τη διεθνή ασφάλεια, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Ονομάζομαι Μπενζαμά Οτκουβιαχτούρ και εργάζομαι στο Ίδρυμα Στρατηγικών Ερευνών των Παρισίων. Μου ζητήθηκε λοιπόν να εκπονήσω μία μελέτη όσον αφορά την ε, διάδοση πυρηνικών όπλων στην Βορειοανατολική Ασία. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα, τα βασικά πορίσματα της μελέτης μου και ελπίζω στη συνέχεια να έχουμε και το χρόνο για να κάνουμε μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για τα ζητήματα αυτά. Χάρη ακριβώς στις παρατηρήσεις σας θα είμαι σε θέση να οριστικοποιήσω την έκθεση αυτή με απότερο στόχο να δημοσιευτεί επισήμως και να μπορέσει να δοθεί και σε άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πυρηνική και βαλιστική κρίση της Βορείου Κορέας είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Ουσιαστικά αποτελεί εξίσωση πολλών διαφορετικών παραμέτρων και μεταβλητών, ορισμένες από τις οποίες είναι ακόμα στάθμητες και άγνωστες σήμερα. Τα αποτελέσματα επίσης των πρόσφατων προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ αποτελούν το νέο αστάθμητο παράγοντα της εξίσωσης αυτής. Θα κάνω λοιπόν κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις όσον αφορά το τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε από τη μελλοντική αμερικανική πολιτική μετά την, μάλλον υπό των πρόσφατων αποτελεσμάτων. Συνοψίζοντας, ή μάλλον, προτού μιλήσουμε για τις πολλές προσπάθειες που έχουν γίνει προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόγραμμα, το βαλιστικό και το πυρηνικό της Βορείου Κορέας, θα ήθελα να σας πω πώς έχουν τα προγράμματα αυτά με τα οποία ασχολείται η διεθνής κοινότητα, για τα οποία ανησυχεί τόσο έντονα. Τι γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτά τα προγράμματα. Ένα πράγμα που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι τα πυρηνικά και παλαιστικά προγράμματα της Βορείου Κορέας έχουν ε, βελτιωθεί με πολύ επικίνδυνο ρυθμό από την αρχή της δεκαετίας μας και από τότε που έφτασε στην εξουσία ο Κιμ Ιονγκ Ουν στις αρχές δηλαδή του 2012. Όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, οι τελευταίες πυρηνικές δοκιμές γίνανε τον Σεπτέμβριο, στις 19 Σεπτεμβρίου και το σύστημα επαλήθευσης της συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών είδε ότι όντως υπήρχαν σεισμικές δονήσεις στην περιοχή αυτή, 5,1 της κλίμακας Ρίχτερ, δονήσεις που οφείλονταν στις δοκιμές αυτές που έκανε η Βόρεια Κορέα. 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ ήταν η δόνηση που, αξιολόγησε, που αξιολόγησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Το εύρος, η, η ακτίνα των δονήσεων αυτών ήταν 15 με 20 χιλιόμετρα και αν συγκρίνουμε τα δεδομένα αυτά με, το με την πρώτη δοκιμή που έγινε στις αρχές του 2016, μπορούμε να πούμε ότι έχει διπλασιαστεί αυτή τη στιγμή η ισχύ σε αυτών των δοκιμών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυξάνεται πάρα πολύ επικίνδυνα ο ρυθμός με τον οποίο γίνονται οι δοκιμές αυτές 2006, 2009, 2013 και 2016 είναι ημερομηνίες και τις οποίες είχαμε τέτοιες δοκιμές. Επί του παρόντος η ικανότητα της Βορείου Κορέας για την παραγωγή πλουτονίου είναι 6 κιλά ετησίως, πράγμα το οποίο αντιστοιχεί σε μία βόμβα σε τήσια βάση. Η χώρα λοιπόν αυτή έχει αρκετά πλουτόνιο αυτή τη στιγμή για να κατασκευάσει 6 με 8 βόμβες, δηλαδή 32 με 54 κιλά πλουτονίου. Διαθέτει αυτή τη στιγμή η Βόρειος Κορέα. Όσον αφορά τώρα την παραγωγή ψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, Σύμφωνα με τον Σίκφριτ Χέκερ, έναν Αμερικανό ερευνητή ο οποίος πήγε σε ένα τέτοιο κέντρο της Βορείου Κορέας το 2010, φαίνεται ότι ε, όντως θα μπορούσε η Βόρεια Κορέα να δημιουργήσει ουράνιο υψηλού βαθμού, ε, ε, ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού 150 κιλά HEU, δηλαδή ποσό που αντιστοιχεί σε 6 περίπου βόμβες και αυτό αντιστοιχεί σε 350 με 400 κιλά όσον αφορά τη μελλοντική παραγωγή δηλαδή της Βορείου Κορέας. Βλέπετε λοιπόν ότι το καθεστώς αυτό έχει το απαραίτητο σχάσιμο υλικό για να φτιάξει 20 με 25 βόμβες μέχρι τα τέλη του 2016. Και αυτό βέβαια εξαρτάται από τις διάφορες εκτιμήσεις που έχουμε. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα πάλι με εκτιμήσεις, 24 με 26 τέτοιες ε, βόμβες δοκιμάστηκαν από το καθεστώς, αποτέλεσαν αντικείμενο δοκιμών, 12 τέτοιες δοκιμές γίνονται το 2015, 19 τέτοιες δοκιμές το 2014 και 7 δοκιμές το 2013. Ο ρυθμός λοιπόν πάλι των βαλιστικών αυτών προγραμμάτων έχει αυξηθεί τόσο πολύ κατά το έτος 2016 που μπορούμε πλέον να κάνουν μια συγκεκριμένη διάκριση ανάμεσα στους επιχειρησιακούς πυράβλους και του πυράβλους που αναπτύσσονται, που βρίσκονται ακόμα σε φάση δοκιμής. Χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή δοκιμές όσον αφορά διάφορες κατηγορίες πυράβλων, όπως η πυράβλη μουσουνταν Μουσουντάν, Σκούντ ή KN11. Και μόνο και μόνο το 2015 έχουν γίνει πολλές δοκιμές και για τις τρεις αυτές κατηγορίες πυράβλων όσον αφορά το νέο πύραυλο KN11 και KN14. Πάλι προβλέπεται εδώ πέρα μία δοκιμή τόσο για τον πύραυλο αυτό όσο και για το σύστημα εκτόξευσής του. Όσον αφορά τον RBM που ονομάζουμε συνήθως πύραυλο Μουσουντάν έχει δοκιμαστεί 9 φορές το 2016. Οι δύο τελευταίες δοκιμές έλαβαν χώρα πριν από δύο εβδομάδες και από ό,τι φαίνεται απέτυχαν. Τι σημαίνει αυτό. Η Βόρειος Κορέας Καταρχάς, δεσμεύεται πάρα πολύ για την ανάπτυξη του πυράβλου αυτού και από ό,τι φαίνεται μπορεί να έχουμε μια επιχειρησιακή συσκευή που σχετίζεται με τον πύραυλο αυτό το 2017 ή το 2018. Οι περισσότεροι τώρα εκτοξευτήρες έχουν να κάνουν με τον πύραυλο Σκούντ. Ο RMB1 πύραυλος, καθώς επίσης και ο K1 02 έχουν δοκιμαστεί, πάλι έχουν γίνει 12 δοκιμές για τους πυράβλους αυτούς σε τίσια βάση. Και αυτό το οποίο φαίνεται να είναι νέο στην όλη ιστορία είναι ότι όλες αυτές οι βαλιστικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας έχουν γίνει αντιληπτές από τη διεθνή κοινότητα. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 2016 η KCNA, η βασική δηλαδή μονάδα ενημέρωσης της Βόρεια Κορέας, είπε ότι θα έκανε δοκιμή μιας, ενός νέου πυράβλου και σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή τύπου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένας νέος εκτοξευτήρας για τον πύραβλο αυτό. Ουσιαστικά καταδεικνύεται κατά αυτόν τον τρόπο ότι η χώρα έχει την απαραίτητη ικανότητα προκειμένου να μπορεί να και να προχωρήσει διαστημικά προγράμματα και να φτιάχνει το απαραίτητο υλικό το οποίο απαιτείται για την εκτόξευση των πυράβλων αυτών. Πρέπει επίσης να πούμε ότι οι δυνατότητες οι στρατιωτικές της Βορείου Κορέας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με υπερβολή, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει δείξει ακόμα η χώρα ότι μπορεί όντως να εκτοξεύσει ένα ICBM. δεν έχει επιδείξει επίσης ότι όντως μπορεί να δημιουργήσει πυρηνικές κεφαλές και ότι θα μπορούσε να τις εξοπτεύσει στην ατμόσφαιρα. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι Ακόμα και αν γίνουν πιο αυστηρέ οι κυρώσει κατά του καθεστώτο τη Βορείου Κορέα, ακόμα και αν υπάρξουν περισσότερε κυρώσει κατά των πυρηνικών και βαλιστικών προγραμμάτων τη Βορείου Κορέα, η χώρα αυτή, από ό,τι φαίνεται, έχει τι δυνατότητε να συνεχίσει τα βαλιστικά αυτά προγράμματα με του δικού τη μονοπόρου. Όσον αφορά την συμμετοχή της Βορείου Κορέας στις δραστηριότητες διάδοσης πυρηνικών όπλων σε παγκόσμιο επίπεδο, πράγμα το οποίο ανησυχεί εξίσου βέβαια τη διεθνή κοινότητα, το καθεστώς αυτό βλέπουμε ότι έχει ήδη κάποιους μηχανισμούς που αρχικά είχαν δημιουργηθεί προκειμένου να μπορεί να προμηθεύεται αγαθά και τεχνολογίες που κανονικά υποτίθεται ότι υπόκεινται σε διεθνείς κανονισμούς. Ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθεί το καθεστώς να χρηματοδοτήσει τα βαλιστικά της προγράμματα προκειμένου να μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητες αυτές διάδοσης πυρηνικών όπλων, μολονότι υπάρχει ένα αυστηρό καθεστώς κυρώσεων κατά της χώρας. Όσον αφορά την διάδοση πυρηνικών όπλων από τη Βόρεια Κορέα, γνωρίζουμε ότι χώρες όπως η Λιβύη ή η Συρία είχαν συνεργαστεί με τη χώρα αυτή χωρίς όμως να υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για τέτοιες συνεργασίες. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ε, απτά δεδομένα. Όσον αφορά την διάδοση βαλιστικών πυράβλων, έχει αποδειχθεί ότι η Πιον Γιάνκ έχει υποστηρίξει το πρόγραμμα παραγωγής όπλων που χρησιμοποιούσε ουράνιο στη Συρία και Υπήρχαν επίσης συμφωνίες συνεργασίας με την Συρία το 2002 και με το Ιράν το 2012. Και σύμφωνα με τους περισσότερους εμπειρογνώμονες και αναφέρομαι σε ορισμένους Αμερικανούς εμπειρογνωμόνους, δεν υπάρχουν πολλά αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι πραγματικά υπήρχε μια συνεργασία μεταξύ των τριών αυτών χωρών όσον αφορά την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων θα πρέπει να δούμε τα πράγματα ήδη από την αρχή της δεκαετίας του 1990. Για να είμαι σύντομο, θα πω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την υφιστάμενη πραγματικότητα. Οι κυρώσεις είναι ο βασικός διπλωματικός δρόμος που είχε χρησιμοποιηθεί για να, σταματήσει, να σταματήσουν τα προγράμματα αυτά στην Βόρειο Κορέα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, από τότε δηλαδή που κατέρευσαν οι εξαμερείς συνομιλίες μετά την άνοιξη δηλαδή του 2007. Αν δούμε ότι ε, επιταχύνεται ο ρυθμός δοκιμών στην Βόρεια Κορέα, Υπάρχουν συγκεκριμένα ψηφίσματα των ΗΕ Εθνών που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σαφώς συμβολικά εφόσον δεν έχουν καταφέρει να ανατρέψουν το ρυθμό αυτών των δοκιμών. Άλλοι θα μπορούσαν να πούνε ότι δεν αναζητήσαμε ως διεθνή κοινότητα εναλλακτικέ λύσεις. Πάντως το καθεστώς των διεθνών κυρώσεων όντως έχει γίνει πιο αυστηρό και πιο σκληρό τελευταία χρόνια, ιδίω μετά την ε, έγκριση του ψηφίσματος 2217 των Ηνωμένων Εθνών το Μάρτιο του 2016. Οι κυρώσεις λοιπόν αυτές είναι αρκετά αμφιλεγόμενες. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ενδεχομένως ακριβώς εκεί πέρα θα έπρεπε να επικεντρωθούμε, ότι αυτό θα πρέπει να απασχολήσει όλους τους εμπλεκόμενους στην αντιμετώπιση αυτή τη κρίση. Το Συμβούλιο Ασφαλεία των Εθνών ενέκρινε πέντε συνολικά ψηφίσματα κατά τη Βορείου Κορέα κατά των προγραμμάτων αυτών από τότε που ξεκίνησαν οι πρώτες υπόγειες δοκιμές το 2006 και κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα διεθνές καθεστώς κυρώσεων κατά της Βορείου Κορέας, όπου ουσιαστικά έχει ως στόχο να μην έχει πρόσβαση πλέον η Βόρειο Κορέας, η Βόρεια Κορέα τελικά που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για τα πυρηνικά της προγράμματα. Μεταξύ του 2006 και του 2013 το διεθνές αυτό καθεστώς κυρώσεων προοδευτικά ενισχύθηκε, αλλά συνδεόταν πάντα σε μία αποδεδειγμένη διασύνδεση μεταξύ των δραστηριοτήτων της Βορείου Κορέας και των προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής. Εκεί ακριβώς είχαν αντιπιστεί κάποια κενά στο πρόγραμμα αυτό των κυρώσεων και μάλιστα ορισμένε από τι διατάξει των ίδιων των ψηφισμάτων αυτών των Ηνωμένων Εθνών ερμηνεύονται διαφορετικά από τη μία χώρα στην άλλη. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε και ποια ήταν η πολιτική βούληση των βασικών εμπορικών εταίρων της Βορείου Κορέας, οι οποίες δεν δείξαν την απαραίτητη βούληση για κυρώσεις κατά της Βορείου Κορέας. Ας μην ξεχνάμε ότι η Κίνα παραδοσιακά αποτελεί σύμμαχο της χώρας αυτής. Γνωρίζετε τα υπόλοιπα στοιχεία όσον αφορά τις κυρίως ένα 17 με 18% της υποστήριξης προς τη Βόρειο Κορέα προέρχεται από την Κίνα. Η Κίνα μάλλον αντιστοιχεί στο 76% του συνολικού εμπορικού όγκου της Βορείου Κορέας και από τα 500 εκατομμύρια δολάρια έχουμε περάσει στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια του 2014 όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Βορείου Κορέας και Κίνας. Επομένως η Κίνα δεν παίζει το παιχνίδι της διεθνής κοινότητας ή παίζει ένα άλλο παιχνίδι. Δεν έχει χρησιμοποιήσει την οικονομία της ως μόχλευση προκειμένου να μειωθεί η επιθετική συμπεριφορά της Βορείου Κορέας το ψήφισμα 2217 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών του Μαρτίου του 2016 έχει τροποποιήσει σαφώς ε, το επίπεδο φιλοδοξίας ε, των Ηνωμένων Εθνών και έχει δημιουργήσει ουσιαστικά ένα πλήρες δεσμευτικό